Okay. Uh, dear colleagues. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Χαίρομαι ιδιαίτερο που καλωσορίζω τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έδειξε προθυμία να έχει αυτή τη συνάντηση μαζί μας. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η χρονική στιγμή γιατί θέλουμε να ενημερωθούμε για την συμφωνία που επετεύχθη τον Ιανουάριο σε σχέση με την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος. Επίσης, χθε συζητήθηκε το θέμα στο Eurogroup. Θέλουμε να δούμε και τις προοπτικές, ε, την προοπτική των συζητήσεων σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους. In light of the... Ε, Κάτι επίσης σημαντικό. Ενώ ολοκλήρωση ε, του προγράμματος. Ο πρόεδρος του Eurogroup χθε έκανε μια δήλωση. Είπε ότι έχουμε εξαιρετικά ναι. Θα ακούσουμε την αξιολόγηση και του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι η τεχνική ομάδα για τα ζητήματα χρέους και ε, οι σχετικές εργασίες θα προχωρήσουν. Θα ακούσουμε τον Ευκλήδη βέβαια. Και οι συνάδελφοι φαντάζομαι ενδιαφέρονται επίσης να δουν πώς προχωρούν τα τα τι γίνεται με τα προαπαιτούμενα. Γενικότερα ποιες είναι οι προοπτικές ε, οικονομικής δραστηριότητας και τι σενάρια μπορούμε να περιμένουμε μετά το τέλος του μνημονίου. Δημόσια συνεδρίαση και δίνω το λόγο στον Υπουργό Τσακαλώτο για να μας κάνει την παρουσίασή του. Σε ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Λιγότεροι ε, είναι οι παρόντες, ε, που σημαίνει μάλλον ότι υπάρχει λιγότερος πανικός ε, και μεγαλύτερη ηρεμία για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Άρα λιγότερο ενδιαφέρονται για την κατάσταση στην Ελλάδα. Προχωρά ε, η κατάσταση, βελτιώνεται όταν θα βγει από το μνημόνιο και όταν θα έχει αλλάξει εντελώ το ρυθμό τη και το βηματισμό τη, η Ελλάδα πιστεύω ότι θα λένε ότι ο Ιούλιος του 2017 και το τότε Eurogroup ήταν το πιο σημαντικό, το πιο κομβικό Eurogroup γιατί τότε επιτεύχθηκε η τελική συμφωνία για το χρέος που βέβαια τις λεπτομέρειες δεν τις έχουν ακόμη συζητήσει όπως είπε ο Ρομπέρτο τώρα ξεκινάει η συζήτηση αλλά οι γενικές γραμμές συζητήθηκαν τότε. Επίσης, ε, στη τελευταία παράγραφο της δήλωσης του Eurogroup ε, του Ιουνίου του 2017 αναφέρεται ότι είναι έτοιμο το Eurogroup να υποστηρίξει την Ελλάδα με περαιτέρω χρηματοδότηση για να δημιουργήσει αυτά τα κεφαλακά μαξιλάρια, αυτά τα ταμιακά αποθέματα. Και αυτό μας ε, επέτρεψε να έχουμε τον Ιούλιο κάτι πολύ μια πολύ επιτυχημένη εξέλιξη, μια πριν τα Χριστούγεννα που ήταν μια ανταλλαγή, αν θέλετε, για να είναι πιο ε, ελκυστικά τα ομόλογα και η τρίτη την προηγούμενη εβδομάδα. Τρεις εξόδους είχαμε στις αγορές και υπό δύσκολες συνθήκες όλα αυτά. Η τρίτη αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί όμως. Ε, υπάρχουν δύο ε, εκρεμή προαπαιτούμενα που κατά κάποιο τρόπο δεν είναι στον έλεγχο της κυβέρνησης. Το πρώτο είναι ότι περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το ελληνικό. Σύντομα την περιμένουμε αυτή την απόφαση. Και το δεύτερο αφορά την συνέχιση των ροών των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήθελε να έχει ε, περισσότερες πληροφορίες προτού λάβει την τελική της απόφαση. Μίλησα με τον Πιέρ Μοσκοβισή και με τον Μάριο Σεντένο, ο οποίος ε, είπε ότι δεν προβλέπει μελλοντικά προβλήματα. Όπως και αν έχει, ήδη ε, έχουμε οργανώσει την επίσκεψη των θεσμών για τις 26 του μήνα. Τετραήμερη επίσκεψη για να ξεκινήσει η διαδικασία για την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση. Και μαζί με αυτό νομίζω ότι στους επόμενους τρεις-τέσσερις μήνες ε, μέχρι τον ε, Ιούνιο που έχουμε Ιουνίου του επόμενο Eurogroup θα συμπληρωθούν τρία-τέσσερα κομμάτια του πάζλ. Ένα είναι η τέταρτη αξιολόγηση, όπως είπαμε. Το δεύτερο κομμάτι του πάζλ είναι το θέμα του χρέους, το οποίο συζητείται τώρα στην ομάδα εργασία του Euro Working Group και κάποια αποτελέσματα θα υποβληθούν στο Eurogroup του Μαρτίου, δεύτερο κομμάτι του πάζλ αυτό. Τρίτο θα είναι η φύση της εξόδου, πόσο κοντά θα είμαστε σε σχέση με Πρωτογαλία, ε, Κύπρο, Ιρλανδία, τι θα γίνει με την ε, εποπτεία μετά την έξοδο από το μνημόνιο, πόσο γρήγορα μπορούμε να ενταχθούμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το καθεξής. Δεν φαντάζομαι ότι περιμένει κανείς μέχρι τις 28 Αυγούστου να έχουν ρυθμιστεί όλα αυτά. Να αποφύγουμε δηλαδή ένα ταπικό ε, Eurogroup που ξεκινάει 3 το μεσημέρι και τελειώνει 3 το πρωί. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι πολύ νωρίτερα, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο. Για να περάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, ως ελληνική κυβέρνηση προσπαθούμε να είμαστε δραστήριοι Κάτι που δεν ήταν εύκολο να είναι κανείς ε, διορατικός και να προγραμματίζει εκ των προτέρων. Γιατί σε ένα πρόγραμμα προσαρμογής υπάρχει μεγάλη πίεση, πας από μια κρίση στην άλλη, προσπαθώντας να λύσεις το τάδε πρόβλημα, το δίνα πρόβλημα. Και ένα από τα μειονεκτήματα του να είναι κάποιο σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι ότι είναι δύσκολο να προγραμματίσει ε, να κάνει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όμως τώρα νομίζω ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό το σχεδιασμό τον Απρίλιο, μετά το Ορθόδοξο Πάσχα, θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ολιστικής ανάπτυξης, τη στρατηγική μας, την αναπτυξιακή μας στρατηγική. Για να δείξουμε και στις αγορές και στους θεσμούς και στα κράτη-μέλη, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Πώς βλέπουμε την περίοδο μετά το μνημόνιο, τι είδους μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν θέλουμε να συνεχιστούν, πώς θα έχουμε μέτρα φιλικά προς την ανάπτυξη και πώς θα συνδυάσουμε με κοινωνικά μέτρα ώστε όλη η κοινωνία να νιώσει ότι συμμετέχει στην επιστροφή στην ανάπτυξη. Δεν θέλουμε δηλαδή εκπλήξεις μετά την περίοδο των μνημονίων. Θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει λίγο πολύ τι προβλέπουμε μέσω πρόθεσμα και σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να προχωρήσουμε. Πολλές, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις εσείς βοηθήσατε πάρα πολύ. Έχετε έρθει στην Ελλάδα, έχω έρθει και εγώ εδώ, αλλά περισσότεροι δεν γνωρίζουν το φάσμα αυτών των μεταρρυθμίσεων που έχει καλύψει πάρα πολλού τομεί. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει από την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής θα έλεγα. Έχουμε κάνει με το κτηματολόγιο πρόοδο, με τη χρήση της γης και της, ε, με τη δόμηση και την ανάπτυξη γενικά. Αυτό βοηθάει και τους επενδυτές. Έχουμε λοιπόν τις βασικές μας προτεραιότητες και υπάρχουν και τα κοινωνικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Εξίσου σημαντικό όμω και για την Ευρώπη. γιατί υπάρχει επιφυλακτικότητα και υπάρχουν αυτές οι φυγότερες δυνάμεις. Είναι ε, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα και αυτή η ανησυχία ότι η Ευρώπη δεν ανήκει ε, στους Έλληνες. Είναι εν μέρει ασφαλμένη εντύπωση αυτή, εν μέρει όμως έχει ένα έρισμα. Um, uh, deficit. So I don't want to give a, a big talk. I thought that I would give the... Δέκα λεπτά είχα στη διάθεσή μου. Θα σταματήσω εδώ για να υπάρξουν να υπάρξει περιθώριο για ερωτήσεις και απαντήσεις. We start with the questions, I guess. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε με τις ερωτήσεις. Στρέφομαι εκ δεξιών μου. Κύριε Κίρτσο, παρακαλώ. And thank you, Minister. Two questions. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχουν να κάνουν με τη... η πρώτη έχει να κάνει με τη συζήτηση που είχατε με τον πρόεδρο Τράγκη στο Eurogroup. Διαβάζω τον ελληνικό τύπο. Υποτίθεται ότι ήταν έντονη, θερμή συζήτηση, δεν ξέρω ακριβώς, και είχε να κάνει με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ε, συζήτηση. Δεν ξέρω ποιους κανόνες μυστικότητας και απορρίτου έχετε στο Eurogroup, αλλά αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη, θα σας ευχαριστούσα πολύ. Και ένα δεύτερο που ενδιαφέρει κυρίως την Ελλάδα. Έχει να κάνει με ορισμένα μέτρα που η κυβέρνηση έχει οθετήσει για τα έτη 2019-2020. Μιλούμε για την μείωση των παλαιότερων συντάξεων που έχουν ήδη δοθεί, χορηγηθεί. Έχετε νέα για αυτό το ζήτημα, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση στους πολιτικούς κύκλους και στην κοινωνία στην Ελλάδα, ότι δηλαδή η Ελλάδα, η κυβέρνηση προσπαθεί να επαναδιαπραγματευτεί αυτά τα μέτρα, γιατί έχουν ένα προφανές κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον για την ίδια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Υπουργός, χθες στο Eurogroup γινόταν μια συζήτηση και για το επταετές ομόλογο το οποίο εξέδωσε η Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα και θεώρησα και πίστευα ότι και ο Κλάους Ρέγκλιν και ο Μάριο Ντράγκη ήταν ίσως υπερβολικά απεσιόδοξοι. Και για να είμαι ειλικρινής, μιλούμε ε, για μια διαφορά στο βαθμό και όχι στο είδος. Είπαν ότι είναι ένα σύστημα προειδοποίησης για το ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε εσφαλμένα. Αλλά εγώ απάντησα ότι ήταν ε, εξαιρετική η επιτυχία με δεδομένες τις πολύ αρνητικές συνθήκες που επικρατούσαν στις διεθνείς χρηματαγορές. Γιατί τη νύχτα που έκλεισε η έκδοση του ομολόγου, ε, ο Dow Jones είχε ε, πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Έγινε μια συζήτηση λοιπόν γι' αυτό σε πολύ φιλικούς όρους και μετά έγινε συζήτηση για το προαπαιτούμενο που περιέγραψα, που ένα από τα δύο προαπαιτούμενα που δεν έχουν ακόμα κλείσει οριστικά. Και Πιστεύω ότι το ζήτημα ήταν το εξής. Τι λέει το προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής, απρόσκοπτης ροής διενέργειας ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Εμείς λοιπόν έχουμε συστήσει, έχουμε συγκροτήσει και έχουμε νομοθετήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις λεπτομέρειες για τη μετάβαση από τους φυσικούς πληστηριασμούς στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Έχουν υποβληθεί ενστάσεις. Κατά την άποψή μου ως κυβέρνηση νομίζω ότι αρκετά έχουμε κάνει ως προς αυτό το θέμα για να κλείσει το προαπαιτούμενο. Έχουν ψηφιστεί όλα αυτά και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν πολύ πιο αυστηρή για αυτό το ζήτημα από ό,τι θα χρειαζόταν. Και αυτό είπα. Ε, έχω, τρέφω μεγάλο σεβασμό με, για το, στο πρόσωπο του Μάριου και νομίζω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Βεβαίως μπορεί να έχουμε αδιαφωνίες στις απόψεις μας για διάφορα ε, ζητήματα και σίγουρα θα υπάρξουν και στο μέλλον. Τώρα, για το θέμα ε, του, των μέτρων και αντίμετρων μετά τη λήξη του προγράμματος, γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα μέτρα που έχουν εγκριθεί για το 2019, έχουν εγκριθεί και αντίμετρα και είναι ένα ε, σύμφωνο, μια δέσμη μέτρων δημοσιονομικός ουδέτερη η οποία προβλέπει κάποιες μειώσεις στις συντάξεις αλλά έχει από την άλλη και μάλιστα για πρώτη φορά στην Ελλάδα προβλέψεις και μέτρα για στήριξη ατόμων χαμηλής και μεσαίας κοινωνικής τάξης και της στέγασής τους είτε είναι ενοικιαστές είτε έχουν δάνειο υποθήκη στο πλαίσιο ενός προγράμματος καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα και γι' αυτό ο δημοσιονομικός αντίκτυπος είναι ουδέτερος. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί δεν υπάρχουν συζητήσεις και είναι πολύ νωρίς να πούμε ε, κατά πόσο όλα αυτά θα είναι μέρος των επικείμενων διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Πολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συζητούμε την έξοδο, αλλά ήταν μια τελείως διαφορετική έξοδος αυτή που συζητούσαμε πριν από δυόμιση χρόνια. Όταν ε, ε, συζητήθηκε η δυνατότητα για μια προσωρινή έξοδο από την Ευρωζώνη. Χαίρομαι που τώρα συζητούμε την έξοδο που είναι επιθυμητή για όλους μας, την έξοδο από το πρόγραμμα για το ελληνικό κράτος και την ελληνική κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ε, καταφέρνει να σταθεί στα πόδια της και το γεγονός ότι επιτρέπουμε στους Έλληνες πολιτικούς επιτρέπεται να κάνουν τα δικά τους λάθη, λέει ο μιλητής. Ε, νομίζω ότι είναι καλό αυτό και είναι καλό το γεγονός ότι η πολύ ψηλή ανεργία σημειώνει μεγάλη μείωση, σημαντική μείωση. Η έξοδος ε, που συζητούμε τώρα είναι όχι μόνο η έξοδος από το πρόγραμμα αλλά και η έξοδος προς τις ε, χρηματαγορές, τις αγορές κεφαλαίων και προς τον... Και αυτό ε, θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα άλλων μελών του Eurogroup. Πρέπει να είναι αξιόπιστη έξοδος και πρέπει να γίνει συζήτηση αυτή για την ελάφρυνση του χρέους. Εγώ είμαι από τις κάτω χώρες και ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση και στις κάτω χώρες και στη Γερμανία. Αλλά το 2010 και το 2012 ήταν προς το συμφέρον ε, της Ολλανδικής και της Γερμανικής αγοράς να υπάρχουν αυτά τα δάνεια για να ενισχυθεί και η αγορά ομολόγων. Επομένως σας ρωτώ για τα θέματα της συζήτησης της ελάφρυνσης χρέους, τι είναι αυτό που ελπίζετε και περιμένετε και από την άλλη για να είναι επιτυχημένη η έξοδος πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη δημοσιονομική οικονομική πολιτική. Ίσως υπάρχει κάποια νευρικότητα εκεί. Πώς σχεδιάζετε να επιτύχετε αυτή την αξιοπιστία αφού με την έξοδο από το πρόγραμμα πρόγραμμα δεν θα μπορείτε να δανείζεστε ε, με το γνωστό τρόπο του προγράμματος και δεν θέλετε και την προληπτική πιστοτική γραμμή από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα θέλετε να ε, πετάξετε με τα δικά σας φτερά είδα την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου από το 3,6 πήγε στο 4,2 ξαφνικά, πολύ γρήγορα, άρα δείχνει ότι επικρατεί νευρικότητα και συνεχίζεται η νευρικότερα στις χρηματαγορές, άρα πρέπει να ενισχυθεί η αξιοπιστία σας για να μην έχουμε εκρήξεις και εκτοξεύσεις στα ομόλογα. Πώς θα πιστεύετε ότι θα τα πετύχετε αυτά. Ο κύριος Υπουργός, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για το θέμα της αξιοπιστίας, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πραγματικά οικοδομήσει, χτίσει πολύ περισσότερη, πολύ μεγάλη αξιοπιστία τα τελευταία δύο-δυόμιση χρόνια και αυτό φαίνεται και στις αγορές, αλλά και στις σχέσεις μας με τα θεσμικά όργανα και με το Eurogroup. Αυτό οφείλεται επίσης και στα γεγονότα και στους αριθμούς. Έχουμε υπεραπόδοση στους δημοσιονομικούς στόχους για τρίτη συνεχή χρονιά και αυτό το μου φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό και γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο. Και παρά τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει οι Έλληνες, τις οποίες καθόλου δεν θέλω να πίσω και ούτε κι εσείς το πράξατε άλλωστε, έχουμε επιστροφή στην ανάπτυξη και η κείμενοι αριθμοί στην ε, οικονομία είναι πολύ δυνατή. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές ε, παρουσιάζουν αριθμητικά στοιχεία εξαιρετικά θετικά και μάλιστα σε κλάδους που δεν θα το φανταζόταν κανείς στην Ελλάδα. Έχουμε ανάπτυξη, ας πούμε, στα μέταλλα, στην ενέργεια, στο λογισμικό, ε, στους, σε αυτούς τους κλάδους παραγωγής. Πράγματα, δηλαδή, πολύ ενθαρρυντικά και αυτός είναι ένας τρόπος ενίσχυσης ε, της ε, αξιοπιστίας μας. Δεν είμαι σίγουρος ότι η προληπτική πιστοτική γραμμή δίνει σε μια χώρα περισσότερη αξιοπιστία. Δεν συμφωνώ με αυτό. Αντεχομένω είναι ένα σήμα προς τις αγορές ότι εμείς δίνουμε στην Ελλάδα προληπτική πιστοτική γραμμή γιατί δεν εμπιστευόμαστε την Ελλάδα και άρα μπορεί να δράσει αυτό με τον αντίθετο τρόπο. Το ε, νόημα κάθε προγράμματος είναι κάποια στιγμή να βγει κανείς από αυτό. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι άλλος ο στόχος, έτσι δεν είναι. Και κάποια στιγμή και νομίζω ότι είναι καλή στιγμή αυτή ε, του Ιουλίου γιατί και η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει και η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει. Είναι λοιπόν μια θετική και ευτυχή συγκυρία να συμβεί η έξοδος ε, στο πρόγραμμα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να πω ότι ατύχησαν λίγο σε σχέση με την έλευση της κρίσης στη χώρα μας και την προόδο και εξέλιξη αν θέλετε της ε, παγκόσμιας κρίσης. Νομίζω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και στην ελληνική κυβέρνηση και υπάρχει εμπιστοσύνη εμπιστοσύνη και στα συνδικάτα και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα ότι θα μπορούσαν όλοι να σταθούν στα πόδια τους και ε, δεν θα χρειάζονται συνέχεια να είναι συνδεδεμένοι ε, με το μηχάνημα, ε, των αναπνευστήρα αν θέλετε. Υπάρχει το ταμιακό απόθεμα, υπάρχει αυτό το μαξιλάρι για να ε, καταλαγιάσει τις αγορές. Δεν μπορεί να έχει κανείς κεφαλαιακό μαξιλάρι από τη μία και προληπτική πιστοτική γραμμή από την άλλη. Δεν έχει νόημα. Έχει κανείς μία ζώνη προστασίας. Πόσες ζώνες προστασίας θα έχει. Έχει μία κουβέρτα να τον προστατεύει. Πόσες κουβέρτες θα, βάλει, ε, θα ρίξει πάνω του. Και τέλος, ε, θεωρώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν ανησυχίες για την Ελλάδα και την ελάφρυνση χρέους. Υπάρχει βεβαιότητα στην αγορά ως προς αυτό, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Δηλαδή τα spread τώρα, οι αποκλήσεις των επιτοκίων ήταν πολύ, είναι τώρα πολύ χαμηλότερα από ό,τι είχε προβλέψει ο οποιοδήποτε μετά την πρώτη έξοδό μας στην αγορές εάν ρωτούσε στην Κομισιόν μετά την πρώτη ε, επιτυχημένη έκδοση ομολόγων πόσο θα ήταν τα spread ε, μετά, ποτέ δεν θα είχε προβλέψει ότι θα ήταν τόσο χαμηλά. Και μάλιστα είχαμε μια μήνυ χρηματιστηριακή κρίση στις ΗΠΑ πρόσφατα. Ε, μετά την, το πρόγραμμα ανταλλαγή ομολόγων είχαμε ένα ράλι πράγματι και ήρθαν ε, οι επενδυτές και τα πούλησαν για να αποκομίσουν τα κέρδη τους. Αυτός είναι και ο σκοπός άλλωστε. Δεν είναι, μας εκπλήσει όταν ε, οι αγορές είναι σε αναταραχή, ότι οι επενδυτές αρχίζουν και πουλούν μαζικά για να εγγράψουν πραγματικά κέρδη. Όμως, ε, όλη αυτή η αξιοπιστία θα κατοχυρωθεί και θα γίνει αντικείμενο εγγύησης μόλις αποκτήσουμε έναν έντιμο, τίμιο συμβιβασμό για το θέμα ε, του χρέους. Μια δέσμευση δηλαδή η οποία θα αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού αναμφισβήτητα και θεωρώ ότι η δουλειά με αυτό το γαλλικό μηχανισμό που έχει συσταθεί και πρέπει να πω ότι εμείς το είχαμε πρωτοσκεφτεί και το είχαμε στην προεκλογική μας εκστρατεία αλλά εν πάση περιπτώσει ένας από τους καθηγητές μου έλεγε δεν έχει σημασία ποιος το είπε πρώτο, σημασία έχει ποιος το είπε τελευταίος και γι' αυτό τώρα αποκαλείται γαλλικός μηχανισμός ρύθμισης τα, ε, για τα, τα του χρέου θέματα. Εν πάση περιπτώσει κλείνω την παρέθμιση για να, παρένθεση για να πω ότι αυτός ο γαλλικός μηχανισμός ε, αυτός ο μηχανισμός δημιουργεί ένα συμβιβασμό για τις πολύ απεσιόδοξες προβλέψεις που έχει το ΔΝΤ για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και αυτό με εκπλήσει γιατί αφού το ΔΝΤ έχει συνεισφέρει τόσο πολύ στα ευρωπαϊκά προγράμματα γιατί είναι τόσο απεσιόδοξο αφού έχει την ε, ευθύνη για πάρα πολλά από αυτά και την υπερβολική αισιοδοξία ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δηλαδή αυτός ο μηχανισμός προσπαθεί να συγκεράσει αυτά τα δύο, την υπεραπεσιόδοξη άποψη του Δουνουτού, την υπεραισιόδοξη ενδεχομένως άποψη των ε, ε, θεσμών και νομίζω ότι έτσι θα καταφέρει να καταλαγιάσει τις ανησυχίες των αγορών. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πρέπει να πάρει κάποια ελάφρυση χρέους και αυτό θα ενισχύσει την αξιοπιστία μας σε μακροπρόθεσμη βάση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Ρομπέρτο. ορίζω και τον κύριο Τσακαλώτο. Δεν υπάρχουν πράγματι πολλοί συναδελφοί εδώ, αλλά κάποιοι υπάρχουμε. Είμαστε εδώ, εγώ μεταξύ άλλων και πρέπει να σας ε, βεβαιώσω ότι ενδιαφέρον για την Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει και για την οικονομική της ε, μοίρα, αν θέλετε. Θα ήθελα να συνεχίσω στον τόνο του Πολ Τάνκ για την αξιόπιστη έξοδο στις ε, κεφαλαγορές μετά την έξοδο της Ελλάδας το τρίτο πρόγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε, ότι δηλαδή αυτή η προληπτική πιστοτική γραμμή θα ήταν σημάδι αδυναμίας προς τις αγορές. Επομένως, αν η Ελλάδα θέλει να είναι αξιόπιστη και θέλει να δείξει ότι είναι ικανή και μπορεί να εξπερτήσει το χρέος της στο μέλλον ε, χωρίς ε, ενίσχυση και μηχανική υποστήριξη, αλλά μόνο στεκόμενη στα δικά τη πόδια, είναι ένα σαφές μήνυμα. Χρειαζόμαστε βοήθεια, όχι. Δεν χρειαζόμαστε γιατί μπορούμε να καταφέρουμε μόνοι μας. Το ερώτημα είναι, στην έκθεση της ΕΚΤ, στην έκθεση του Κοινοβουλίου, για την έκθεση της ΕΚΤ, ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο πρόσφατα, ζητά το Κοινοβούλιο από την να αγοράσει ελληνικό κρατικό χρέος μετά την έξοδο της Ελλάδας από το τρίτο πρόγραμμα. Το ερώτημά μου προς εσάς είναι, εσείς και η κυβέρνησή σας είστε διατεθειμένοι δημοσίως να ζητήσετε από την ΕΚΤ να μην αγοράσει ελληνικά ομόλογα σε κανένα από τα προγράμματα, ώστε να δοθεί στην Ελλάδα η δυνατότητα να καταδείξει ότι είναι ικανή και ισχυρή αρκετά για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα και με αξιόπιστο τρόπο το χρέος της. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα το ερώτημά σας. Αν κατάλαβα καλά θα απαντήσω και αν δεν κατάλαβα μπορείτε να επανέλθετε. Δύο θέματα έχουμε εδώ. σε ό,τι αφορά την αγορά ομολόγω από την έκτο, Το πρώτο είναι η ποσοτική χαλάρωση και το δεύτερο είναι το λεγόμενο waiver. Το πρώτο θέμα που αφορά την ποσοτική χαλάρωση είναι ότι η ΕΚΤ έχει την άποψη, πώς να το ότι θα μπούμε εκεί μόνο αν θεωρηθεί βιώσιμο από την ΕΚΤ το χρέος μας. Δεν έχει κάνει όμως προς το παρόν τη δική της ε, ανάλυση βιωσιμότητας χρέους. Το θέμα είναι να δούμε τι λέει το ΔΝΤ ε, στη δική του ανάλυση μετά και το γαλλικό μηχανισμό που συζητήσαμε πριν θα μπορούσε ανάλογα με το τι λέει το ΔΝΤ να υπάρχει ε, και το ενδεχόμενο, το περιθώριο να μπει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό, θα ήταν ένα καλό σημάδι και θα έπρεπε να το κάνει κατά την απόψή μου, αλλά είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εμένα, δεν μπορώ να το ζητήσω, εξαρτάται από αυτούς, είναι ανεξαρτητό όργανο, αυτόνομο. Δεν νομίζω όμως ότι είναι κρίσιμη σημασία για το πρόγραμμα. Είμαι αισιόδοξο ότι ακόμα και χωρίς ποσοτική χαλάρωση ότι μπορούμε να εξέλθουμε από το πρόγραμμα και το ίδιο ισχύει για το waiver, την εξαίρεση. Δηλαδή, έχουμε τώρα, επειδή είμαστε σε πρόγραμμα, υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Επειδή δεν αποδίδουν τα ομόλογά μας, έχουμε αυτό το waiver και η ΕΚΤ μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα ομόλογα. Όταν όμως πάψουμε να είμαστε στο πρόγραμμα. Βέβαια, ε, ο Φίτς μας αναβάθμισε πρόσφατα, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο επενδύσεων. Τι θα κάνει τότε η ΕΚΤΑ. Και πάλι, νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα για τις ε, τράπεζες με δεδομένη την κατάσταση ε, στην τραπεζική αγορά, το να μην υπάρχει αυτή η εξαίρεση και το να μην αγοράζει ελληνικά ομόλογα μέχρι να φτάσουν στο βαθμό ε, επενδύσεων, που αποφέρουν δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα αλλά ε, δεν είναι τόσο πολύ σοβαρό που να μας αποδυναμώνει. Δηλαδή δεν είναι λόγος για να ζητήσουμε. Είναι δυσανάλογο, για να το πω έτσι είναι δυσανάλογο να ζητήσουμε απλά και μόνο για το waiver αυτό μια προληπτική πιστοτική γραμμή. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα ώστε να χρειάζεται προληπτική πιστοτική γραμμή. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, έτσι επαναλαμβάνω. Έτσι ερμήνευσα εγώ αυτά που είπατε. Το κάνατε πιο πολύπλοκο, λέει ο κύριος Λούκε με την απάντησή σας. Δεν ξέρω αν μπορείτε ίσως να αναδιτυπώσετε. Εγώ θα σας πω ξανά το ερώτημά μου. Λέω, αγορά ομολόγων από την ΕΚΤΑ σε οποιοδήποτε πρόγραμμα PSPP, οποιοδήποτε άλλο από κεντρική τράπεζα, στην αγορά πώς θα τα δουν θα τα δουν σαν ε, μέτρα μηχανικής υποστήριξης αν θέλετε της Ελλάδας που στους επενδυτές θα δείξει ότι χρειάζεται η Ελλάδα τέτοιου είδους υποστήριξη εσείς λοιπόν ή η ελληνική κυβέρνηση είστε έτοιμοι να πείτε όχι δεν τα θέλουμε, μην αγοράσετε το ομόλογά μας σας παρακαλώ. Ακόμη και αν έχουν αυτό το βαθμό για ε, ε επενδυτικά. Δεν θα πήγαινα τόσο μακριά λίγο και τσακαλώτος. Ε. Δεν είναι τόσο άσπρο ή μαύρο η επιλογή που έχουμε να κάνουμε. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι θα ήταν καλό να τα έχουμε, αλλά θα ήταν και καταστροφή να μην τα έχουμε. Πρόεδρος, μιλάμε και για την ποσοτική χαλάρωση που αφορά όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Δεν είναι κάτι πρόσθετο. Ναι, Ρομπέρτο, το ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λούκη. Ναι, δεν μπορώ να πω, θέλω πιο ε, αυστηρούς όρους για να δείξω ότι είμαι ε, αξιόπιστος σε σχέση με τα άλλα κράτη ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Greek, so Θα μιλήσω ελληνικά, οπότε παρακαλώ να βάλετε ακουστικά. Καλωσορίζω τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για τα stress test στα οποία θα επιβληθούν οι ελληνικές τράπεζες. Είναι μια διαδικασία που ξεκινά σε λίγο και θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, την εκτίμησή σου Ευκλήδη για το αν θεωρείς ότι εκεί υπάρχει ένας πιθανός κίνδυνος ε, στην ε, ομαλή εξέλιξη και στην ομαλή πορεία της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα και από τα μνημόνια. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό το δίδυμο πακέτο συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυσης του χρέους σε εφαρμογή όσων ήδη έχουν αποφασιστεί από το Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017 και ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ελληνικής κατασκευής και ιδιοκτησίας το οποίο θα ετοιμαστεί έγκαιρα και το οποίο θα δεσμεύει τη χώρα για, τα, για την περίοδο μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Θα ήθελα γύρω από αυτά τα θέματα αν μπορείς να μας δώσεις περισσότερη ε, μια σαφέστερη εικόνα για το χρονοδιάγραμμα. Έχω υπόψη μου χθεσινές δηλώσεις του Μπρούνο Λεμέρ που λένε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφους του χρέους όπως καταρχήν αποφασίστηκαν στο Eurogroup τον Ιούνιο και ο Μάριος Σεντένο λέει έχουν αρχίσει ήδη τεχνικές συζητήσεις. Θεωρείς ε, δυνατό σε αυτό να υπάρχει μια ε, ολοκλήρωση ε, και πότε. Και το δεύτερο, πότε θα είναι η ελληνική κυβέρνηση έτοιμη να παρουσιάσει αυτό το ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ε, μετά την έξοδο από τα μνημόνια προκειμένου να εγγυηθεί και να πείσει όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη του Eurogroup, τους δανειστές, ότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια εμείς θα διατηρήσουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά και θα θεραπεύσουμε τις παθογένειες που έφεραν τη χρεοκοπία και τα μνημόνια και ε, με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Για πότε βλέπεις να είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα και να εγκριθεί. Σε ό,τι αφορά την ελληνική στρατηγική για την ανάπτυξη, υποσχεθήκαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη στρατηγική μέχρι τον Απρίλιο, μετά το Ορθόδοξο Πάσχα, που είναι μία εβδομάδα μετά το Καθολικό. Οπότε φαντάζομαι θα συζητηθεί στη συνέχεια και στο Eurogroup. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε. Η ιδέα είναι, μάλλον δύο ιδέες. Πρώτον, δέσμευση να μην γυρίσουμε στο μοντέλο του 2008 και πριν. Το μοντέλο προκρίσης δηλαδή. Για προφανείς λόγους. Κάτι πολύ στραβό αυτό το μοντέλο, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Και εσείς δεν θα με καλούσατε να έρθω εδώ. Δεύτερον, όχι απλά δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό το μοντέλο, αλλά θέλουμε και ένα ολιστικό μοντέλο. Δηλαδή το άθροισμα υπερβαίνει, μάλλον το σύνολο υπερβαίνει το απλό άθροισμα των μερών. Αυτό είναι η αρχή που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Και αυτό μπορεί να βασιστεί σε κάποιες ιδέες ίσως για την ενέργεια και άλλους σημαντικούς τομείς όπως ο τουρισμός ή ε, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αλλά όχι μόνο. Θα πρέπει να δούμε η Ελλάδα τι είδου χώρα είναι. Είναι μια χώρα που έχει πάρα πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει και πολλή γεωργία. Άρα, τι θα πει ολιστικό. πώ ταιριάζουν όλα αυτά μεταξύ τους. Όχι μόνο η βασική τομή τα μεγάλα project, αλλά πώ οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν και αυτέ σε αυτά τα μεγάλα project. Είτε είναι ενεργειακά, είτε αφορούν τι μεταφορές, είτε συνδρομικά δίκτυα, λιμάνια, οδικές μεταφορέ και το καθεξής. και πώς καταλήγεις στο τι χρειάζεσαι μετά. Αρκούν τα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία, από την ΕΤΕΠ, τι είδους χρηματοδότηση χρειάζεται, χρειάζεται κάποια παραπάνω χρηματοδότηση, τι σχέση έχει αυτό με την εκπαίδευση, με το είδος του εργατικού δυναμικού, ε, την απασχόληση, την επαγγελματική κατάσταση κτλ. Αυτή είναι μία πτυχή λοιπόν αυτών προσπαθούμε να πετύχουμε και θα μας δείξει τι ε, μεταρρυθμίσεις έχουμε ήδη κάνει. Σας είπα για το κτηματολόγιο, για την έγκριση, ε, για τις φοροαποφυγή. Για να τονωθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να συναρμολογηθούν μεταξύ τους και να δείξουν σε ένα εντελώς νέο μοντέλο. Και αυτό είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν θα καθίσουμε και θα πούμε μια μέρα πώς μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Ήδη το κάνουμε. Παλιά είχαμε τα μεγάλα project, μεγάλα, μεγάλα έργα υποδομών. Ήταν 20% η συμμετοχή των μικρομεσαίων. Τώρα θέλουμε να το αντιστρέψουμε. 80% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 20% μεγάλα project. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο αυτό και τελείως διαφορετικό είδος διακυβέρνησης. Γιατί δεν γίνεται με μια πελατειακή πολιτική και με παρεμβάσεις, αλλά με μια δέσμη κανόνων. Απολύτως διαφανής. Όλοι γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα έργα, πώς μπορούν να υποβάλουν ψηφιότητα και δεν χρειάζεται να πάρουν τον Ευκλήδη, το Γιάννη, τη Μαρία, τηλέφωνο κτλ. κτλ. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, Νομίζουμε ότι κοντεύουμε στην ε, έναρξη της συζήτησης για το χρέος. Στις επιτροπές που συζητούν αυτά τα ζητήματα συχνά δεν καλείται η Ελλάδα να συμμετάσχει και το λέω για να μην λέω πάντα καλά πράγματα, αλλά να ασκήσω και κάποια κριτική. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι και ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ότι δηλαδή γίνονται συζητήσεις για το ελληνικό χρέος στι οποίες δεν συμμετέχει η Ελλάδα και κατόπιν εορτή μόνο στο Eurogroup. Όχι, δεν είναι αυτό ο σωστός τρόπος λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτή είναι μια κριτική απέναντι στο πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κατημέλια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βέβαια, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συζητήσουμε και για τα μεσοπρόθεσμα και για το γαλλικό μηχανισμό. Θα ήμασταν πολύ πιο κοντά, πως είναι προφανές, αν η γερμανική κυβέρνηση ε, είχε συγκροτηθεί πολύ νωρίτερα. Δεν σας λέω κάτι που δεν το περιμένετε, τα ακούσετε φαντάζομαι. Και ελπίζω ότι άπαξ και ε, συγκροτηθεί η νέα γερμανική κυβέρνηση θα επιταχυνθεί ο ρυθμός. Και όχι βέβαια για το πρόγραμμα το ελληνικό, για την έξοδο, αλλά και για σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις που έχουν να κάνουν την Τραπεζική Ένωση, ε, που έχουν να κάνουν το κατά πόσο χρειαζόμαστε, δημοσιονομική ικανότητα, ο σταθεροποιητή για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Τάμι κτλ. κτλ. Υπάρχει ένα όλο θεματολόγιο. Εμείς οι Νοτιοευρωπαίοι ξέρετε πάρα πολύ αποτελεσματικοί και του συνασπισμού του κάνουμε ε, στο pitch φιτίλ. Δεν μα χρειάζονται τόσε μέρε ή εβδομάδε που χρειάζονται οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί. Τέλο πάντων. Για τις δοκιμέ αντοχή στα stress test, ε, για να δώσω μια ειλικρινή απάντηση, Δημήτρη, στην ερώτησή σου, δεν το γνωρίζω και δεν το γνωρίζει και κανείς. Ούτε ο Μάριο Ντράγκη ότι το γνωρίζει. Δεν είναι ζήτημα του ΕΚΤ, της ΕΚΤ, συγγνώμη, ε, δεν μπορεί να το ξέρει. Εγώ πάντως ε, κοιμάμαι καλύτερα σε σχέση με πριν από ένα μήνα. Οπότε είχαν, είχαν ανακοινωθεί κάποια ε, σημεία ανάπτυξης που ήταν ένα κακό σενάριο. Εγώ δυσκολεύομαι να δω γιατί θα έχουν οι ελληνικές τράπεζες πρόβλημα με αυτές τις υποθέσεις και εκτιμήσεις όταν το 2015 ήταν πολύ χειρότερα ε, τα στοιχεία των προβλέψεων. Αλλά η ειλικρινή απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι δεν γνωρίζω. Και νομίζω ότι όταν κάποιο δεν ξέρει κάτι πρέπει να το λέει, πρέπει να το παραδέχεται. Ο κύριος Ούρτασον. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι ένας από τους τομείς που έχουν σημειωθεί βελτιώσεις είναι ο τομέας της φορολογίας και θα ήθελα να σας θέσω ορισμένες ερωτήσεις για αυτό το ζήτημα γιατί τα μέτρα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Έχουμε αυτή τη βάση δεδομένων που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε την φορολογία εισοδήματος και τις κεφαλαιακές ροές. Το πρόγραμμα εθελούσιας αποκάλυψης εισοδημάτων με δυνατότητα ενός είδους αμνηστίας αν τα έχω καταλάβει καλά. Και ασυλίας μάλλον, και ε, δημοσιοποίηση των μεγάλων φοροφιλετών ε, θα θέλαμε να μας πείτε κάποια αξιολόγηση, να μας εκφράσετε την άποψή σας. Όλα αυτά επηρέασαν θετικά την ενίσχυση των εσόδων από τη φορολογία. Είδα τα πρόσφατα στοιχεία και παρόλο που υπάρχει θετική αύξηση, θετικό πρόσημο στα έσοδα από τη φορολογία, υπάρχει σημαντική μείωση από την άμεση φορολογία, από τους άμεσους φόρους. Ένα δις λιγότερο άμεση φόροι εισπράττονται και θέλω να ξέρω τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Ε, με θετικό πρόσωπο πρόσημο λοιπόν έχουμε αύξηση εσόδων φορολογικών, αλλά κάποιου, κάποια έσοδα από κάποιους φόρους έχουν μειωθεί και θα θέλουμε να μάθουμε το λόγο. Ο κύριος Υπουργός, θα ξεκινήσω προσπαθώντας να είμαι απολύτως έντιμος και ειλικρινής. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής ή καταπολέμηση για παράδειγμα της λαθρεμπορίας πετρελαίου ή καπνικών προϊόντων ήταν πολύ πιο δύσκολη τελικά από ότι εμείς ως αριστερά πιστεύαμε ότι θα ήταν. Πιστεύαμε ότι ήταν ένα πολύ πιο εύκολο πρόβλημα να λυθεί από ό,τι τελικά αποδείχθηκε ότι είναι. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα κινούνται και έχουν κινηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζουμε υπεραπόδοση, υπερεπιδότηση επιδόσεις ε, στα έσοδα, γιατί όλα αυτά δεν τα μετρούν οι θεσμοί ως συνεισφέροντα ε, για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων γιατί τα αποκαλούν μη παραμετρικά μέτρα. Τα παραμετρικά μέτρα είναι μόνιμη αύξηση ας πούμε στο φορολογικό συντελεστή που θα ισχύσει για πάντα. Η αύξηση σε συγκεκριμένο συντελεστή ε, ΦΠΑ είναι μόνιμη και μπορεί να ε, συνυπολογίζεται πάντοτε και γι' αυτό θεωρείται παραμετρικό μέτρο. Ενώ μια ενίσχυση στα φορολογικά έσοδα μπορεί να είναι παροδική θεωρούν οι θεσμοί και γι' αυτό αποκαλείται μη παραμετρικό ε, μέτρο. Και ο λόγος για τον οποίο ε, τα αντιμετωπίζουμε είναι ε, ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε είναι να έχουμε τέτοιες πολιτικές, να ενισχύσουμε το σύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών και αυτό έχει βοηθήσει ιδιαίτερο στο να συλλέγεται περισσότερος ΦΠΑ. Οι διασταυρώσεις είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και είμαι πολύ περήφανος διότι στο Υπουργείο μου ε, ε, δημιουργήθηκε αυτό το λογισμικό το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο. 15 με 20 άνθρωποι εργάζονταν για ένα ολόκληρο χρόνο, χωρίς αργίες, χωρίς Σαββατοκύριακα. Ε, φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Τι να σας πω. Ε, να σας πω ότι διασταυρώνουμε τις καταθέσεις των ατόμων στις τράπεζες με προηγούμενες ε, δηλώσεις τους φορολογικές. Δηλαδή, ο Ρομπέρτο έχει ένα εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα και έχει όλες οι δηλώσεις του την τελευταία δεκαετία είναι ότι έχει έσοδα ετήσια 10.000 ευρώ. Τώρα, μπορεί αυτό να εξηγείται διαφορετικά, αλλά είναι ένα καμπανάκι που σημαίνει συναγερμό για να ελέγξουμε τον Ρομπέρτο ακόμα περισσότερο. Τρόπος του λέγει. Φαίνεται εύκολο. Πόσο δύσκολο να είναι θα μπορούσα να έχω ένα τραπεζικό λογαριασμό με ένα εκατομμύριο ευρώ σε μια ελληνική τράπεζα και μετά να το πάρω, να το κάνω έμβασμα σε μια άλλη ελληνική, να το βάλω μετά την άλλη μέρα στην τρίτη ελληνική και μετά την τέταρτη μέρα να το στείλω στην BNP ή στην Deutsche Bank. Άρα πρέπει να εντοπίζεται ένας μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που δεν τον έχει κανείς άλλος. Και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο, γιατί ε, για να μην θεωρηθεί ότι ο Ρομπέρτο έχει 4 εκατομμύρια από 1 εκατομμύριο σε κάθε τράπεζα και σε κάθε λογαριασμό που τηρεί. Το πρόβλημα δηλαδή ήταν αυτό, είναι πιο περίπλοκο από ό,τι ακούγεται. Και αυτό έχει να κάνει με το καρότο και το ε, μαστίγιο οι θεσμοί δεν μας επέτρεψαν να έχουμε περισσότερη ασυλία και αμνηστία όσοι είχαν οι Ιταλοί στην εθελούσια αποκάλυψη εισόδεμάτων. Ε, ε, δηλαδή πληρώνεις αυτά που θα πλήρωνες αν είχες αφήσει τα χρήματα στην Ελλάδα χωρίς πρόστιμα. Αυτό ήταν το ε, καρότο που δώσαμε στον κόσμο για την εθελούσια αποκάλυψη των εισόδημάτων. Να σας πω το εξής το να ανακαλύψει ένας υπάλληλο ότι κάτι πάει λάθος με ένα συγκεκριμένο φορολογούμενο ή ε, φορολογικό μητρό χρειαζόταν 8 με 9 μήνες στο παρελθόν και τώρα χρειάζεται 5, μήνες, 5 λεπτά το, ο υπάλληλο να το ανακαλύψει. Έχουμε δηλαδή συντμίσει τους χρόνους. Είναι πολύ δύσκολο να συντμίσουμε τους, τους χρόνους για τον έλεγχο στη συνέχεια. Ένα τυχές γεγονός είναι το ότι δεν τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά σε ένα ζήτημα, διότι τα δικαστήρια αποφάσισαν ότι παλαιότερες υποθέσεις πρέπει να παραγραφούν και δεν μπορούμε να ερευνήσουμε για ε, φοροδιαφυγή παλαιότερων ετών. Αυτό ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό για εμάς. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι νομικοί λόγοι, αλλά ε, θεωρητικά θεωρείται ότι όσο πιο παλιά είναι η υπόθεση φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής που συναντάς και ερευνάς, τόσο χαμηλότερη είναι η φοροαποφυγης που συναντας και ερευνας τοσο χαμηλοτερη ειναι η εισπραξιμοτητα αν ε, τελικά καταφέρεις να δικαιωθείς ως δημόσια αρχή. Και υπάρχει και το θέμα των μεγαλοφιλετών και της δημόσιας αποκάλυψης των ονομάτων τους. Ε, ένα συγκεκριμένο τμήμα, το ΚΕΦΟΜΕΠΑ, ασχολείται με αυτό και το τελευταίο χρόνο έχουμε διπλασιάσει τα εισοδήματα τα έσοδα που έχουμε από 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ίσπραξη φορολογικών χρωστουμένων από μεγαλοφιλέτες, έχουμε φτάσει στα 700 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε διπλασιάσει δηλαδή τις επιδόσεις μας σε ό,τι αφορά την εισπραξιμότητα από μεγάλους φοροφιλέτες. Είπα στην αρχή ότι οι θεσμοί δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα μη παραμετρικά μέτρα, τις μη παραμετρικές μεθόδους και έχουν ε, προβλέψει με πολύ μικρή απόδοση τα μέτρα αυτά. Έχουν πολύ χαμηλές προβλέψεις και γι' αυτό ζητούν ε, αυξήσεις των φόρων που δεν ήταν απαραίτητες επειδή θεωρούσαν ότι ε, θα είχαν χαμηλή απόδοση τα μέτρα αυτά και τελικά δεν την είχαν. Ε, ένα αρνητικό αποτέλεσμα ήταν για το ε, φόρο εισοδήματος και για τις συνεισφορές ε, τις εργασιακές ε, στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αυτό, σε αυτό οφείλεται η μείωση των εσόδων από τους άμεσους φόρους τις οποίες αναφερθήκατε, γιατί οι θεσμοί ε, προβλέπουν ότι η απόδοση των μέτρων θα είναι χαμελότερη από αυτό που αποδείχθηκε ότι ήταν τελικά και ε, γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη τους τα μη παραμετρικά μέτρα. Έχουμε 3,5 δις φορολογικές περικοπές τα επόμενα χρόνια και αυτό θα είναι σημαντικό. Τώρα, υπάρχει ένα δίλημα για κάθε υπουργό. Όταν εντοπίζει κάτι, το αλλάζει αμέσως το αλλάζει αμέσω ναι για να διορθώσει ένα σφάλμα. Αλλά απ' την άλλη αν το αλλάζει αμέσω, δίνει το μήνυμα ότι κάθε τρει και λίγο αλλάζει η φορολογία, αλλάζει η νομοθεσία για τη φορολογία και αυτό δημιουργεί νευρικότητα. Θέλουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις ξαφνικής μείωσης κατά ένα δις ευρώ ας πούμε του ε, φόρου που συλλέγεται από τους άμεσους φόρους των εσόδων του κράτους. Δεν θέλουμε δηλαδή κάθε έξι μήνες να υπάρχει μια αλλαγή. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι από αυτά που με ρωτήσατε. Ευχαριστούμε κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ναι, θα τα πω στα γερμανικά, βάλτε τα ακουστικά. Ήταν η Επιτροπή Ελεγχού του Υπερπολογισμού στην Αθήνα και στη Λέσο την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα απλά να σας πω ότι πραγματικά υπήρχαν ε, τα ε, πάρα πολλά προαπαιτούμενα και είδαμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ε, βελτιώσεις ό,τι αφορά το κτηματολόγιο όπως είπατε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που όλα τα μέτρα ε, τα οποία είχαμε όλοι συστήσει, τα 180 κτλ. έχουν αποδώσει αποτελέσματα και θα είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο κράτος Ελλάδα με πολύ σύγχρονη διοίκηση. Το πρώτο μου ερώτημα σε σχέση με τη διοίκηση, ε, το η κρατική υπάλληλη που ήταν το 4% των ε, ασφαλισμένων και ήταν πολύ επιβαρημένο το ασφαλιστικό σύστημα λόγω αυτού. Τι σχέδιο υπάρχει τώρα, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κόστος. Ε, πρέπει να αλλάξει κάτι σε αυτό, γίνονται κάποιες προσπάθειες και σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκεται σε τι ε, κατάσταση και επίσης να μας πείτε πού μπορούμε να σας υποστηρίξουμε, πού πιστεύετε ότι μας χρειάζεστε και μπορούμε να συνεισφέρουμε. Αυτά και κατά τα άλλα καλή επιτυχία και συγχαρητήρια μέχρι τώρα. Thank you very much. I'm not sure I captured the first... Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα το πρώτο σας ερώτημα για τη δημόσια διοίκηση. Ναι, το μεγάλο ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων ήταν το ερώτημα που επιβαρύνει τη κοινωνική ασφάλεια. 30% είναι το ποσοστό. Τι σχέδια έχει η κυβέρνηση. Θα αλλάξει αυτό το ποσοστό. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το μόνιμο τεράστιο κόστος. Um, so you'll... Oh, no, I don't need that, do I? Uh, <laughs> um, um, so you'll allow me to answer your... Αν επιτρέπετε να απαντήσω αργότερα στο πρώτο σας ερώτημα. Εξακολουθώ να μην είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει τι εννοείται με το 30%. Δεν ξέρω, δεν μου στέλνετε καλύτερα ένα email και μέσω του Ρομπέρτ, γιατί το είχαμε ξανακάνει την τελευταία φορά. Υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις που δεν ε, τις κατήχα εντελώς και μου έστειλε ένα email ο Ρομπέρτο και απάντησα. Να συζητήσω λοιπόν πρώτα τα περί ιδιωτικοποιήσεων και το τι ε, βοήθεια θα μπορούσε να μας προσφερθεί από πλευρά σας και αφού σας ευχαριστήσω βέβαια για τα πολύ καλά ευγενικά σας λόγια σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποίησεις. Ε, υπάρχουν δύο πτυχές ε, στο μέτωπο της αποκρατικοποίησης. Η πτυχή πρώτη αφορά το πρόγραμμα των αποκρατικοποίησεων και επίτα υπάρχει και το ζήτημα του ε, Ταμείο Επενδύσεων. Ε, άρα και στα δύο μέτωπα έχουμε πρόοδο ό,τι αφορά τις ε, ιδιωτικοποίησεις οποίες ήταν όριμες. Έχουμε αυτό το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, Αποκρατικοποιήσεων. Περιμένουμε η ΔΕΣΦΑ, η Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, το ελληνικό πάει πιο γρήγορα, Περιμένουμε λοιπόν τη ΔΕΣΦΑ και υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδιωτικοποίησεις που προχωρούν και προσπαθούμε να βρούμε ενδιαφέροντες τρόπους ε, για να ε, υπάρχει αμοιβαίο όφελος και για τους πιστωτές αλλά και για εμάς. Το άλλο μέτωπο έχει να κάνει τα... με τα περιουσιακά στοιχεία και τις κρατικές επιχειρήσεις, με τα ακίνητα. Εκεί δεν έχουμε μόνο το μέτρο των ιδιωτικοποιήσεων για να έχουμε περισσότερη αξία. Υπάρχει η ιδιωτικοποίηση, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, μακροχρόνιες μισθώσεις, ε, κάποιες κοινοπραξίες και άλλα μέτρα που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Έχουμε την Εποπτική Επιτροπή και το Σχετικό Φορέα, το Δικτικό Συμβούλιο και θα ξεκινήσει αξιολόγηση σύντομα. Για να δούμε την ποιότητα αυτών των ακινήτων. Θέλουμε να έχουμε ποιοτικές επενδύσεις ε, και για τις ε, μισθώσεις ε, και για τα ακίνητα. Υπάρχουν πολλά ελληνικά ακίνητα που θα μπορούσε κανείς να να πάει στις αγορές και να αυξήσει ε, την αξία τους και τα κέρδη να μοιραστούν μεταξύ κράτους, δημοσίου, ε, πιστωτών ε, και επενδυτών. Αυτά στο πλαίσιο και της αναπτυξιακής στρατηγικής, για την οποία μίλησε και ο κύριος Παπαδημούλης. Έχουμε λοιπόν την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας που έχει αναλάβει το θέμα αυτό. Για το τρίτο σας ερώτημα, πού, μπορούμε να, πού μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε. Μιλάτε αυστηρός για τη δική σας επιτροπή ή γενικότερα για την Ευρώπη, για τα κράτη-μέλη, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η δική σας επιτροπή πρέπει να πω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και η επιρροή της ήταν σημαντική. Το ίδιο και η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, ήταν μια διαφορετική φωνή, αν θέλετε, σε σχέση με το σε επιδόσεις της Ελλάδας. Έχουμε τώρα διάφορα ζητήματα που είναι υποσυζήτηση, όπως το ενδεχόμενο ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμού. Και νομίζω ότι εδώ η ελληνική εμπειρία μπορεί να είναι πολύτιμη. Έχει κανείς να διδαχθεί πολλά. Ε, είπα ήδη ότι υπάρχουν συζητήσεις για το ελληνικό χρέος στις οποίες δεν παρίσταται η Ελλάδα, δεν είναι καν προσκεκλημένη. Μπορούμε να συζητήσουμε τα ελεγκτικού συνεδρίου που υπήρχε ένα είδος μικροδιαχείρισης που δεν θεωρώ ότι βοήθησε και ε, θα μπορούσε να είναι καλύτερη η αντιμετώπιση και η σχετική νομοθεσία. Επομένως, καλό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει πιο ισχυρή φωνή ε, για να έχουμε στο δυνατόν ε, μια πιο καθαρή έξοδο και ελάφρυνση του χρέους. Βέβαια, το θέμα ε, είναι και πάλι εδώ η ανάπτυξη. Υπάρχει μια συζήτηση, φαντάζομαι θα συμμετέχει και η δική σας επιτροπή, μια συζήτηση στην Ευρώπη για το κατά πόσον χρειάζεται η λεγόμενη δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρώπη, το fiscal capacity, για να δημιουργηθεί ενέδωση σταθεροποίηση. Έχουμε το γαλλικό μηχανισμό επενδύσεων, οι Ιταλοί προτείνουν κάτι διαφορετικό μια ασφάλιση ανεργίας κτλ. Ξέρω ότι οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Σκανδιναβοί θεωρούν ότι υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Δεν υπάρχει όμως ε, ηθικός κίνδυνος στις ε, πολιτικές σταθεροποίησεις, γιατί ουσιαστικά ε, μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό των απολειών. Δηλαδή αν χάνει ένα ε, ε, δολάριο ε, η Ομοσπονδιακή, λέω για τη ΣΥΠΑ, Αν χάνει Federal, το υποστηρίζει 12-13 σέντ και όχι παραπάνω. Το θέμα είναι να μην είμαστε μονίμως ασθενείς και να, ζητούμε συνεχώς ενίσχυση από τη Γερμανία, την Ολλανδία, από τις σκανδιναβικές χώρες. Και το θέμα εδώ, επαναλαμβάνω, είναι η ανάπτυξη και όχι η σταθεροποίηση. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Πολιτική θα πρέπει να δουν προς το μέλλον τι γίνεται. Υπάρχει και η ατζέντα Μακρόν-Μέρκελ. Αυτά τα οποία συζητούνται πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει τρία πόδια. Το ένα είναι η ανάπτυξη ε, και πώς επιτυχάνεται η σύγκληση. Το δεύτερο πόδι είναι τα κοινωνικά θέματα τι θα γίνει με την εργατική τάξη, με τη μεσαία τάξη. Και το τρίτο πόδι, που είναι και το τελευταίο πάνω στο οποίο μπορείτε να βοηθήσετε, είναι η διαφάνεια και η δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Οποιαδήποτε αλλαγή προέρχεται από την ανάγκη μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης και της Ευρώπης να οδηγεί σε μεγαλύτερη λογοδοσία και μεγαλύτερη δημοκρατία, διότι πώς να το πω, οι Ευρωπαίοι δεν είναι απλά επιφυλακτικοί και διστακτική για την Ευρώπη επειδή ε, δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική ευαισθητοποίηση, αλλά και γιατί δεν υπάρχει αίσθηση του ανήκειν. Δηλαδή νιώθουν ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τι αποφάσει που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, μπορεί να βοηθηθεί με την εμπειρία και την τεχνογνωσία, να δημιουργηθούν, ε, δηλαδή να καταρτιστούν έργα ε, αναπτυξιακά, ποιοτικά τι λείπει στην Ελλάδα τελικά, χρηματοδότηση ή καλά έργα. Μπορεί κανεί να το συζητήσει. Για μένα λείπουν και τα δύο. Αλλά δεν ε, λείπει μόνο η χρηματοδότηση, αυτό είναι το σίγουρο. Υπάρχουν ε, πολλέ χώρε στι οποίε δεν υπάρχουν πολλά καλά έργα ε, με την οικονομική απόδοση επιστροφή. Άρα είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να έχουν μια προσέγγιση που θα βοηθήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία, τέτοια έργα δηλαδή να προωθούν. Η ικανότητα δημιουργίας, κατάρτισης έργων ποιοτικών είναι το σημαντικό. Thank you very much. We have concluded our time and uh, I think uh, we had... Uh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ευκλήδη Στακαλώτο, όχι μόνο για την πολύ καλή σας εμφάνιση, τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις, αλλά και την πολύ καλή σας δουλειά, η οποία ήταν βασικό στοιχείο για να επανέλθει η Ελλάδα στην ανάκαψη και για να παρουσιάσει ε, υπερβολικές επιδόσεις, εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, στον τομέα της διαχείρισης, της διακυβέρνησης, της κοινωνικής ε, δικαιοσύνης για την κοινωνικώς δίκαια ανάληψη του βάρους για τις πολιτικές υπέρ του, της ανάπτυξης. Πολλά μένει να γίνουν και συμφωνώ μαζί σας. Ένα από τα βασικά στοιχεία για την αξιοπιστία είναι ότι η δική σας πλευρά είναι αξιόπιστη, ε, ε, ολοκληρώνει και υλοποιεί πλήρως την ατζέντα και θα πρέπει να υπάρξει επαρκές επίπεδο ελάφρυσης χρέους και είναι κάτι που μπορούμε να, στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε και ελπίζω μετά τις 4 Μαρτίου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καθέσουν στο τραπέζι για να οριστικοποιηθεί και αυτό το θετικό σημείο. Και άλλωστε στην Επιτροπή μας η, η δίκαιη πρόσβαση πρέπει η δίκαιη πρόσβαση σε αυτή την Επιτροπή όπου θα συζητηθούν τα θέματα του χρέους όλων είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Άλλωστε, μιλούμε για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα, αλλά μιλούμε και για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ζώνη του ευρώ θα αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτού του περίπλοκου και παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη συνοχή με πιο δημοκρατικό, πιο διαφανή τρόπο θα προσπαθήσουμε όλοι να συμβάλλουμε προς αυτή τη διαδικασία και θα συνεχίσουμε και το διάλογο με εσάς και με όλους όσοι ε, θα εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα στο μέλλον. Ευχαριστώ.